Welcome back uh, to the committee meeting. Um, I have to inform. στην συνεδρίασή μας και πάλι. Μου είπαν ότι δεν θα έχουμε προς τα σλοβακικά διερμηνία σήμερα το, πρωί. Και επίσης να σας ε, υπενθυμίσω ότι 9 με 10 και μισή σήμερα έχουμε την κυρία Μωρά Σατζή, η οποία έχει καλέσει κάποιους συμπατριώτες της από την εκλογική της περιφέρεια. Δεν ξέρω αν ήρθαν. Αν ήρθαν πάντως καλώς όρισαν. Όσον αυτές τις τριμερές διαλόγους και τη, στατιστικά για, τα, την κοινωνική πολιτική και το σχετικό σχέδιο οικονομισμού είχαμε τη δεύτερο τριμερή διάλογο. 26 ε, Απριλίου έγινε και έχει σημειωθεί αξιολογή πρόοδος σε τεχνικό επίπεδο ε, ήταν η συνάντηση, αλλά έχουμε και στις 16 Μαΐου αυτή τη βδομάδα το απόγευμα μια συνάντηση τώρα όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων ε, από τα μεταλλαξιγόνα και τα καρκινογόνα, το δεύτερο πακέτο. Έχουμε τον πρώτο τριμερή διάλογο. Ο κύριος Ζωλά είναι ο εισηγητής. Και από αυτού θα έχουμε τριμερή διάλογο αυτή τη βδομάδα στις 17 Μαΐου το πρωί. Επίσης, χθες το απόγευμα, λίγοι ήμασταν εδώ, αλλά είχαμε καλέσει κάποιους ε, ε, ερευνητές, κάποιους ειδικού για ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση. Και πώς επηρεάζεται ο επαγγελματικό βίος, ο κοινωνικό βίος από ε, αυτά τα φαινόμενα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση μεταξύ τους και ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον μια που ήμασταν τόσο λίγοι και θα πρέπει να σας πω ότι έτσι ενστικτοδός θεωρώ ότι θα μας ξανάρθει αυτό το θέμα και σύντομα κιόλας. Γιατί έχουμε πολλά σοβαρά σχετικά ζητήματα τα οποία απαιτούν, επιβάλλουν μια συζήτηση εις βάθος. Οπότε, όσοι ήταν χτες εδώ το απόγευμα θα χαρούν γιατί θα επανέλθουν. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια θα έχουμε και ε, καινούργια πρόσωπα να έρθουν να μας τα πούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για τη συζήτηση αυτή, για τις επιπτώσεις ε, με των μέσο άνθρωπο ε, και τον πραγματικό του βίο στο άμεσο μέλλον. Πέραν αυτόν τώρα. Προχωρούμε. Έχουμε το σημερινό σημείο υπαριθμών 1. Είναι το έκτο στη συνολική τη διάταξη όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτικής ζωή για του γονεί και του φροντιστέ. Έχουμε ε, 660 τρόπο πέραν των 80 του εισηγητή. Επομένως, έγινε πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά και ευθύς αμέσως να δώσω στον εισηγητή τον λόγο. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, όπως τα είπατε. Ήταν πολύ θετικό νομίζω όλο αυτό το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το θέμα μου. Καλά, δεν έχουν έρθει και πολλοί βουλευτέ σήμερα το πρωί, αλλά το ενδιαφέρον το καταδεικνύουν όλε αυτέ οι τροπολογίε. Η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ε, κινούνται στο ίδιο μήκο κύματο. Και να μην αναλώνουμε το χρόνο μα για αυτά στα οποία συμφωνούμε. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, όμως που αναδεικνύουν αντίθετες θέσεις και επίσης ε, οι περισσότεροι πάντως από τους συναδέλφους συμφωνούν στο εξής. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να θεωρηθούν τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να υπάρχουν υπηρεσίες φροντίδας και επίσης θα πρέπει να πλαισιώσουμε τους αναπήρους και επίσης όχι μόνο σε γέννηση αλλά και σε υιοθεσία, αν προβλέπεται πατρική άδεια, επίσης να χορηγείται σχετική άδεια, να υπάρχει αύξηση του ποσού που δεν επιδέχεται μεταβίβαση όσον αφορά την, ε, την πατρική άδεια για τους φωτιστές πέντε ημέρες και επίσης Επίση ε, να ρυθμιστεί το θέμα του ποιο και πότε ε, ζητεί την πατρική ή μητρική άδεια σχέση με την ηλικία του παιδιού. Οπότε έχουμε διάφορα σημεία. Όμως που υπάρχουν κάποιες τριβές, κάποιες διαφορές θα πρέπει να ζητηθούν γιατί έχουν υποβληθεί και τροπολογίες μεταξύ των δύο άκρων του ναι και του όχι. Επίσης έχουμε διάφορες προτάσεις για πλήρη μισθό σε όλες τις περιπτώσεις ούτως ώστε ε, τελικά όμως να είναι αυτό εθνική αρμοδιότητα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει το, θέμα της, ε, ε, της, του επιδόματος σε περίπτωση ασθενείας θα πρέπει να ρυθμιστεί και θα πρέπει να βασιστεί στον ακαθάριστο μισθό. Επίσης έχουμε τις τροπολογίες των κρατών μελών και πάνε από 45% και φτάνουν στο 100% σε σχέση με αυτού του είδους το επίδομα, σε σχέση με το ανακαθάριστο μισθό. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις διάφορες ε, άδειε που έχουν ε, προταθεί. 8 με 12 έτη το παιδί για την πατρική άδεια και σύμφωνα με την εντύπωσή μου είναι ότι αυτοί που είναι υπέρ της, ε, της αύξησης στο 12 και κάποιοι άλλοι θέλουν να μείνει το όριο ηλικίας παιδιού στα 8 να το συζητήσουμε. Πάντως το 10 είναι ένας συμβιβασμός, να τον πάμε στις διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Τέλος πάντων, να δούμε σήμερα πώς θα τα πάμε στη συζήτηση τώρα όσον αφορά τον ορισμό. Το τι θα γίνει με την άδεια για αυτούς που παρέχουν φροντίδες. Να δούμε τι γίνεται με τους συγγενείς και ποιος είναι ο ορισμός του συγγενούς. Να το συζητήσουμε και κατέληξουμε σε κάποιο συμβασμό. Τώρα όσον αφορά την υποχρεωτικότητα της πατρικής άδεια. Τι να σας πω, δεν είμαι σίγουρος τι θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Να πούμε σε αιτιολογική παράγραφο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, να την ε, θεσπίσουν ως υποχρεωτική την πατρική άδεια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν υπάρχει αναλογικότητα στην ε, οδηγία επ' αυτού. Πάντως ε, ευχαριστώ να το συζητήσουμε τις μέσα επόμενες μέρες. Όσον αφορά την ρύθμιση για την γονική άδεια, για τις μονογονικές οικογένειες διάφορα αναφέρθηκαν και προσπάθησα να αυξήσω τα δικαιώματα των γονέων σε μονογονική οικογένεια, να αυξηθεί αυτή η άδεια. Θα είμαστε στις προσπάθειες, στις τροπολογίες για να υπάρχει ισορροπία και τα μέτρα να μην χαρακτηρίζονται από υπερβολικότητα. ε, να μην καταντήσουμε αυτό να αντικίνητρο για το να προσλάβει ο εργοδότης ε, κάποιον που είναι γονέας μονογονικής οικογένειας. Οπότε θα πρέπει επίσης να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να μην υπάρχει δυσαναλογία και για να είναι επιτυχής μια νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να υπάρχει κάποια ρήτρα διαφύλαξης. Έχουμε σχετικά κάποιες τροπολογίες σε σχέση με το πρώτο σχέδιο κειμένου. Έτσι νομίζω ότι περιφρουρούνται τα συμφέροντα εργοδοτών και μιμιέψεων Οπότε είναι κατακλείδη ολοκληρώνει τη δουλειά για τον πρώτο γύρο εξέταση των τροπολογιών. Σε πολλά συμφωνούμε, θα τα πούμε με τους πιο ηγητές σε επόμενες μέρες και θα τα πούμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο συμφωνούμε και σήμερα θα συνεδριάσουμε και αύριο και ξέρω ότι το Συμβούλιο κινείται προς την κατεύθυνση του να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη από όσα έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ένα προβληματάκι. Πάντως, αυτό επιβάλλει εμείς να έχουμε σώροπη αντιμετώπιση, να είμαστε λογικοί. Οπότε ευχαρίστω και να συνεχίσω την συνεργασία με τους ε, συναδέλφους της Επιτροπής μας και αισιοδοξώ θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία εδώ στο Κοινοβούλιο και δεν είναι τόσο πολύ για το αν θα τα βρούμε εδώ μεταξύ μας. Το θέμα τι θα κάνουμε στον τριμέρι Άρα να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και να καταλήξουμε σε κάποια ισορροπημένη ε, έκθεση ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο γιατί εκεί θα αναδειχθούν τα προβλήματα πολύ περισσότερο από όσα συνάντησα εδώ με τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε το λόγο στους σοσιαλιστές και δημοκράτες και την σκιώδη τους Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά υπάρχει αλληλεπικάλυψη των επιτροπών και έτσι δεν είναι εύκολο να είμαστε, μάλλον αδύνατο να είμαστε παντού την ίδια στιγμή. Άκουσα την, ε, μάλλον δεν πρόλαβα να ακούσω την ε, παρέμβαση του εισηγητή, αλλά τα έχουμε συζητήσει και ξέρουμε ότι σε πολλά σημεία συμφωνούμε και ε, μπορούμε να πούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι καλή που σίγουρα χρειάζει περαιτέρω τροποποιήσεων, τροπολογιών, όμως γενικά καλύπτει τους τρεις στόχους που θέλουμε εμείς να υπερασπιστούμε ως σοσιαλιστές και δημοκράτες, αλλά ξέρω ότι και ο κύριος Κάζα έχει ακριβώς ε, τις ε, ίδιες ε, σκέψεις. Πρώτον, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Δεύτερον, τα μέσα που μπορούμε να δώσουμε για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας. Εδώ οι απολαβές είναι σημαντικές. Και τρίτον, η καταπολέμηση των στερεοτύπων. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ε, προωθήσουμε αυτή την έννοια, την της ε, μη δυνατότητας μεταφοράς του δικαιώματος για να αναθεωρήσουμε τα στερεότυπα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά του, τις ανδρικές και γυναικές δουλειές, αν θέλετε, και το ρόλο του στην οικογένεια. Σε ό,τι αφορά την πρόταση που καλύπτει αυτούς τους τρεις στόχους, θεωρώ ότι παρόλα αυτά μπορούμε κάποια πράγματα να τα βελτιώσουμε στην πρόταση. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την πατρική άδεια, νομίζω ότι θα ήταν καλό αυτή η πατρική άδεια να γίνει υποχρεωτική. Γιατί βλέπουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όταν υπάρχει δικαίωμα στην πατρική άδεια, που υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή, αυτό δεν σημαίνει ότι το αξιοποιεί ο εργαζόμενος, γιατί υπάρχει ο παραδοσιακός ρόλος ε, του άντρα και ε, επικρίνεται εάν ε, αξιοποιήσει αυτό το δικαίωμα. Οπότε πρέπει να πούμε ότι η πατρική άδεια δεν είναι δικαίωμα, αλλά υποχρέωση. Και έτσι θα καταφέρουμε να αυξήσουμε την αξιοποίηση αυτού του δικαιώματος από τους άνδρες. Δεύτερον, να λάβουμε υπόψη την πατρική άδεια ακόμα και όταν ε, το παιδί χάνει τη ζωή του κατά τη γέννηση συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει το δικαίωμα στην πατρική άδεια. Νομίζω ότι και ο πατέρας και η μητέρα έχουν το δικαίωμα να θρηνήσουν ε, το παιδί που χάνουν κατά τη γέννα. Και νομίζω λοιπόν θα πρέπει να χορηγείται αυτό το δικαίωμα στην πατρική άδεια και σε αυτή την περίπτωση και αυτό να αναφέρεται στο κείμενο. Τρίτον, η πατρική άδεια θα πρέπει να δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους και στους αυτοαπασχολούμενους και θα υποβάλουμε τροπολογία υπό αυτή την έννοια. Προτείνουμε επίσης τροπολογία για να υπάρξει ρήτρα μη υπαναχώρησης. Όπως είπα προηγουμένως υπάρχουν πολλά που έχουν ήδη γίνει από τα κρατη Υπάρχει πρόοδος λοιπόν σε πολλά Δεν θα πρέπει λοιπόν με το νέο κείμενο τα ε, κράτη-μέλη να πάνε ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτά που έχουν σήμερα για να ευθυγραμμιστούν με μία οδηγία. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αυτή η ρήτρα της μη επαναχώρησης. Και αυτό που μου φαίνεται το πιο λεπτό σημείο και σίγουρα θα συζητηθεί με το Συμβούλιο είναι το θέμα ε, των απολαβών. Η Επιτροπή αναφέρει έναν κανόνα, ε, η αποζημίωση αυτή, οι απολαβές, να ευθυγραμμιστούν με την ε, άδεια ασθενείας. Αναφέρεται ότι τα ότι η κατάσταση στα κράτη-μέλη διαφέρει πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Ε, προτείνεται από την άλλη για την πατρική άδεια να πάμε στο 75% να διατηρηθεί ε, το σύκλι, δηλαδή η άδεια ασθενεία ε, για την πατρική άδεια. Η δική μας πρόταση θα ήταν να γίνει η ευθυγράμμιση στο 85% του μεικτού μισθού για το σύνολο των αδειών. Ξέρουμε ότι αυτό θα είναι δύσκολο για το Συμβούλιο. Θα είναι μία λοιπόν από τις δυσκολίες για τις οποίες θα πρέπει να δείξουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το ζήτημα ε, του μισθού και των αποζημιώσεων αυτών είναι πολύ σημαντικό. Ιδάλλως θα φτωχοποιήσουμε αυτές τις οικογένειες Γιατί τελικά δεν γίνεται να δίνουμε μία άδεια, αλλά να οδηγεί σε φτωχοποίηση στην οικογένεια επειδή ε, κάνει παιδί. Πρέπει να δώσουμε τα μέσα ε, σε μια οικογένεια που έχει κάνει ένα παιδί και για την οικογένεια αλλά και για την ευημερία του παιδιού. Γιατί βλέπουμε ότι όταν τα παιδιά γεννιούνται σε μια φτωχή οικογένεια, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Τα φτωχά παιδιά είναι αυτά που δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν στην κοινωνία. Οπότε είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα ως προς ε, την ευμερία των παιδιών στην Ευρώπη σήμερα, ιδίως ό,τι φορά τις φτωχές οικογένειες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά είναι συντομία από πλευράς ε, της δικής μας πολιτικής ομάδας. Είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος, γιατί συμμεριζόμαστε αυτές τις αξίες και τις αρχές και θα συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα. Ε, από πλευράς ε, χρονοδιαγράμματος, Ξέρω ότι θα γίνει Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ τον Ιούνιο για το ζήτημα αυτό του timing. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να ακολουθήσει και ε, το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής και του Συμβουλίου για να προσπαθήσουμε και να καταφέρουμε να έχουμε μια πρόταση των σημαντικών δυνατόν. Γιατί περνάει ο χρόνος, ε, σύντομα θα φτάσουμε και στο τέλος της κυριοβουλευτικής θητείας. Καλό θα ήταν λοιπόν να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Προς όφελός μας θα ήταν αυτό και ε, θα καταφέρουμε να έχουμε μια πρόταση που αποτελεί τμήμα της, του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρικε νομίζω ε, αντικαθιστά τη συνάδελφό του που δεν είναι παρούσα εκ μέρου της κυρίας Σινάνσκα που κάπου βρίσκεται, έρχεται προς το Κοινοβούλιο, καθοδόν είναι. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τις, ε, τη βασική της θέση και τι προτεραιότητε τη για τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις. Δεν νομίζω ότι ε, θα κομίζαμε γλάφκα στι Αθήνα αναφέροντας ότι η έκθεση του, των κυρίων Κάζα και καλός ε, αναφέρει ότι οφείλουμε να παραμείνουμε λογικοί όσον αφορά τα αιτήματά μας, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή βάση για τις ε, μελλοντικέ διαπραγματεύσεις σε τριμερούς διαλόγου. Εμείς ε, πρεσβεύουμε τα εξής. Πρώτον, πρέπει η οδηγία να παραμείνει όσο πιο απλή γίνεται. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η οδηγία έχει ως στόχο να καθορίσει ελάχιστα κριτήρια, τα οποία βεβαίως τα κράτη-μέλη θα μπορούν περαιτέρω να διευκρινίσουν. Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να μην γίνει μάχη για τις λεπτομέρειες της πρότασης, καλύτερα αυτό να κρυθεί σε επίπεδο κρατών μελών. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετό περιθώριο έτσι ώστε οι διατάξεις να προσαρμοστούν στις τις ανάγκες που μπορούν να διαφοροποιούνται στα κράτη-μέλη. Δεύτερον, στηρίζουμε την πρόταση του κυρίου Κάζα, ο οποίος ε, υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια υποδομή για τη φροντίδα για τα παιδιά. Και αυτό συμβαδίζει με όλες τις προτάσεις που έχουν σχέση με τις ανάγκες των οικογενειών και την αγορά εργασίας. Τρίτον, για αυτήν την οδηγία δεν θέλουμε αυτή η οδηγία να αποτελεί απειλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εμεί στηρίζουμε ένα κείμενο το οποίο δεν θα έχει ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά στο θέμα της ιδιαίτερης σημασίας για την σκιώδη μας εισηγήτρια, αυτό που παίζει ρόλο είναι η κατάσταση όσων παρέχουν φροντίδα. Θέλουμε να γίνει κάποια αλλαγή στη γλώσσα που χρησιμοποιεί η Κομισιόν στην αρχική διατύπωση. Θέλουμε όμως επίσης να βελτιώσουμε τη θέση των παρεχόντων φροντίδα, να υπάρχει μια ισορροπία έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να έχει το περιθώριο να επεξεργαστεί τα κριτήρια θεωρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε κοινά στοιχεία που μας ενώνουν με την άποψη του κυρίου Κάζα και θεωρούμε ότι οι στόχοι της πρότασης είναι πολύ σημαντικοί για την βελτίωση της ζωής των οικογενειών. Προσβλέπουμε στη συζήτηση και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς κύριε Γκέρικε, οι φιλελεύθεροι έχουν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Βίμπερ. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να εκφράσω την υποστήριξή μου για την άποψη του εισηγητή, για την ε, έκθεση του, ε, της ε, τρόπολογίας που έχει καταθέσει. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κάζα ότι πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές για το τι μπορούμε να επιτύχουμε. Και πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι αυτή η οδηγία να έχει προχωρήσει πριν από το τέλος της θητείας του αυτού του κοινοβουλίου. Γιατί αν δεν το κάνουμε φοβάμαι ότι θα απογοητεύσουμε πάρα πολλούς οι οποίοι θεωρούν ότι η οδηγία αυτή αποτελεί μία ρήξη με το παρελθόν. Δεν είναι ότι θα έχουμε μια ανοιχτή ένα θαύμα, αλλά θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός και πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, βλέπουμε ότι υπάρχει στεναρή αντίδραση στο Συμβούλιο. Άρα δηλαδή θα πρέπει σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου να επιτύχουμε ευρεία και αμέριστη υποστήριξη κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Ε, υπάρχουν πολλές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και εγώ κατέθεσα κάποιες ε, τροπολογίες κυρίως έχοντας κατά νου ότι πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την οδηγία διάφορα είδη εργαζομένων. Οι ε, κατοίκων εργαζόμενοι, αυτοί που εργάζονται κατά πέτηση, αλλά και οι επιτιδευματίες. Επίσης, ε, έχω κάνει και μία ιδιαίτερη σημείωση σχετικά με τις μονογονεϊκές οικογένειες που θα πρέπει να απολάβουν των ίδιων δικαιωμάτων την ίδια προστασία να διασφαλιστεί αυτό στην οδηγία. Επίσης, ε, ορισμός του πατέρα του παρέχοντος φροντίδες ε, για τους τελευταίους ε, πιστεύω ότι είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν σε αυτή την κατηγορία και εργαζόμενοι που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την οικογένεια, οι οποίοι όμως εργάζονται εθελοντικά ε, χωρίς προσπορισμό κέρδους, ε, βεβαίως και με κάποιες εγγύσεις για να ε, μην καθίστανται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Επίσης, να ορίσουμε το τι είναι συγγενής. Πέρα από όλα αυτά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι επίσης να προσφέρουμε στους παρέχοντες φροντίδα ότι εφόσον βρίσκονται σε κράτη-μέλη στο οποίο ισχύουν υψηλέ προδιαγραφές, αυτέ οι προδιαγραφές να συνεχίσουν να ισχύουν και στο μέλλον. Κατά τα άλλα, Μιλάμε για ελάχιστες προδιαγραφές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως ε, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτές οι προδιαγραφές να μην είναι πολύ χαμηλά. Να είμαστε επίσης συνεπείς, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για την κινητικότητα των εργαζομένων, να μπορούν οι εργαζόμενοι να φύγουν από την πατρίδα τους και να πάνε σε μια άλλη χώρα, γνωρίζοντας όμως τα δικαιώματά τους αυτοί που θα μεταβούν. Όπως είπε και ο εισηγητής, ο κύριος ε, Κάζα, σε κάποια θέματα δεν είμαι σίγουρη πόσο πολύ μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά αυτό θα διευκρινιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και πρέπει να σας πω, προσβλέπω σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις που θα συζητήσουμε τους συμβιβασμούς, ε, γιατί αλλιώς χωρίς συμβιβασμούς, αν δεν ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, απλά ε, θα προκύψει εφιάλτης. Μπορείτε λοιπόν να βασιστείτε σε μένα και στο ότι η ομάδα μου θα είναι ρεαλιστική, θα ακολουθήσει μια ρεαλιστική στάση όσον αφορά αυτό το θέμα. κυρία Γκονζάλες Πένιας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως διαπιστώσαμε, έχουμε πάνω από 600 τροπολογίες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από όλες τις πολιτικές πτέρυγες. Να βελτιώσουμε το κύμα, το κάνουμε όσο γίνεται πιο στεγανό. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά με τις τροπολογίες συγκεκριμενοποιούμε αυτά που θέλουμε να διορθώσουμε. Εμείς έχουμε κατεβάσει προς ξαφή κατεύθυνση κάποιες τροπολίες, δηλαδή πώς θα θωρακίσουμε τα, τα ε, συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, να κατοχυρωθεί η θέση της γυναίκας και να υπάρχει όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας ε, συνυπευθυνότητα και έτσι με κάποια μέτρα να ε, πλαισιώσουμε την ε, άδεια επαντρότητας και επίσης να υπάρχει ένα δίκαιο επίδομα δίας τα πιο σημαντικά σημεία να υπάρχει 100% κάλυψη και θέλουμε αυτό του είδους η αμοιβή, αυτό το επίδομα να έχει σχέση με τον μισθό για τους άνδρες. Επίσης υποχρεωτικότητα ε, ημερών και για τους ε, άντρες όπως έχουν οι γυναίκες. Αυτό νομίζω ότι είναι επιθυμητό και δίκαιο. Τώρα όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας έχουμε και κάποιες τροπολογίες ούτως ώστε η... Ε, εκεί που λέμε για την άδεια να λέμε ότι αυτό αφορά εργαζομένους που παρέχουν βοήθειες έτσι να διατυπωθεί σε σχέση τώρα με το, τι ήδη. Ε, προβλέπεται, δηλαδή αυτούς που προφέρουν τύπος κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι δηλαδή που κάθονται στο σπίτι και προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς ε, αμοιβή, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και κάποιους εργαζομένους που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, αλλά με την ε, οδηγία αυτή τώρα θα μπορούν για συγκεκριμένες υπηρεσίες να έχουν συγκεκριμένη ε, άδεια. 12 μέρες ε, το χρόνο, όπως έλεγε η έκθεση ε, των επιπτώσεων. Τώρα όσον αφορά την ευελιξία στην εργασία, θέλουμε αυτό που προβλέπεται να προστατεύει, να ρυθμίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα και επίσης να προσαρμόζονται σαν και των εργαζομένων ε, τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Είναι πιο περίπλοκο αυτό, αλλά νομίζουμε ότι είναι καλύτερο από αυτά τα οποία προβλέπει το σχέδιο οδηγία. Επίσης, θα πρέπει να καλύψουμε τους ε, αυτονόμους, ανεξαρτήτου ε, εργαζομένου που δεν καλύπτονται ακόμη, που δεν κάνουν τις τυπικές μου μορφέ και να καλύψουμε επίσης τους συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού, συγγενείας εξαίματος ή εξαγχιστίας, να καλύψουμε τις ε, οικογένειες ε, τεροφιλοφίλων και ομοφίλων και επίσης θα πρέπει να υπάρχει πλήρης μισθολογική κάλυψη τώρα και ένα νέο στοιχείο είναι το ότι ο εργοδότης μπορεί να απορρίψει την αίτηση άδεια μόνο μια φορά και το πολύ για τρεις μήνες. Τώρα όσον αφορά την ρύθμιση ε, το, το σχετικό με την άδεια αυτό θα πρέπει να κατοχυρωθεί και θα πρέπει εγγράφως να υπάρχει η, η αίτηση και η απάντηση στην αίτηση για να προστατευτούν και εργοδότες και εργαζόμενοι. Να δούμε τώρα το πώς θα αναγνωριστούν στην οδηγία τα συνδικάτα και ο ρόλος τους και επίσης θα πρέπει να προβλέπεται η αναθεώρηση της οδηγίας για την μητρική άδεια και αυτό να γίνει σε τρία ε, χρόνια ούτω ώστε να υπάρξει μια νομοθέτηση για γονική άδεια μητρότητος, και επίση να υπάρχει πλήρης κάλυψη οικονομική, μισθολογική ε, όλων των ε, αδειών. Αυτά όλα μας να ρυθμιστούν και όχι χωριστά στο μέλλον. Και αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα σε τρία χρόνια ούτω ώστε να υπάρχει μόνο μία δέσμη ε, νομοθετικών μέτρων και θα πρέπει τα, η ρύθμιση να σας πιο απλή. και να υπάρχει ενημέρωση για το τι άδειες προβλέπονται. Συμφωνούμε με το ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο για υπαναχώρηση από τα όσα συμφωνήθουν. Άρα, Ελπίζω να συμφωνήσουμε και να στείλουμε μήνυμα ενότητας εν των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους μητροφάνους. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα, γενικώς. να σας πω μια πρατήση και να σας πω για την τροπολογία μας. Αύριο θα τα συζητήσουμε και να δούμε τα κρατημέλη κατά πόσο θα προχωρήσουν προς θέσεις της νομοθεσίες επί τη βάση της πολιτικής που έχουν χαράξει και να δούμε εάν θα πρέπει να προτείνουμε κάποια νέα πρότυπα ως Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και βασικά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί εμείς είμαστε ένα από τα λίγα διεθνή βήματα που για αυτά τα θέματα και την κοινωνική πολιτική δηλαδή νομοθετεί για το καλύτερο. Θα πρέπει να προτείνουμε υψηλά πρότυπα. Αλλά να δούμε εάν θα βελτιωθεί η εθνική κοινωνική πολιτική. Αμφιβάλλω για πολλούς λόγους που αφορούν το πολιτικό ή Πάντως, με τέτοια υψηλά πρότυπα να δούμε πώς θα τάξουμε κάποιους στόχους που μπορεί να απορρίψει το Συμβούλιο ή μπορεί να διαφωνήσει από αυτόν η Επιτροπή, αλλά στο μέλλον αυτοί οι στόχοι θα μπορούν να υλοποιηθούν από την εθνική νομοθεσία. Επομένως, γι' αυτό θα δείτε από πλευράς μας ριζοσπαστικές τροπολογίες. και έχω υποβάλει τροπολογίες για πρώτη φορά ε, είναι η παριθμόν 15. Και λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν για το πώς θα προστατεύσουν τους εργαζομένους σε σχέση με το πώς θα υπάρξει ισορροπία οικογενειακής ζωής και επαγγελματικής ζωής. Άρα τα κράτη-μέλη θα μπορούν να νομοθετήσουν επί τη βάση των διαβουλεύσεων ή επιθεωρήσεων όπως λέμε, σε κάποια κράτη-μέλη. Να ενημερώσουν τα κράτη-μέλη τους εργαζομένους για το πώς μπορούν να πετύχουν περισσότερη ισορροπία επαγγελματικού και οικογενειακού βίου επί τη βάση του ισχύοντος ε, δικαίου, εθνικού δικαίου. και κάποιοι νέοι και φιλόδοξοι του ιδιωτικού τομέα ή του δημόσιου τομέα δεν ξέρουν τι δυνατότητες προβλέπονται για κάποιο είδου κοινωνικά επιδόματα ή για διάφορες ε, άδειε που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Την ισχύουσα νομοθεσία. Βέβαια, θα υπάρξει και κοινοτική νομοθεσία. Και το κράτος επιπληρωμένως θα πρέπει να ενημερώσει αυτούς που ενδιαφέρονται, αυτούς που τους αφορούν αυτές οι άδειες, αυτές οι δυνατότητες που προσφέρονται. Να ενημερωθούν οι οικογένειες, σε σχέση με τις φροντίδες προς τα παιδιά τους. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και άλλες πολιτικές ομάδες. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα αναφέρω τον κατάλογο ομιλητών για να σας καθησυχάσω. Ε, it's Lope Fontanier, it's Moran Chati and it's Jongerius on the list. Gericke, you want to have a... be back on the list. Έλεγε πρόεδρος ότι ο κύριο Γκέριγκε έχει ήδη πάρει το λόγο, αλλά ο ίδιο λέει όχι, μίλησε εξ ονόματο συναδέλφου. Μάλιστα σα βάζω στον ε, κατάλογο μελετών. Από το EFTD. E Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κάζα για την πρόταση που κατέθεσε. Είναι λοιπόν ε, σαφές ότι οι βάσεις αυτής της ε, διαπραγμάτευσης ε, δεν θα πρέπει να είναι προς τα κάτω. Και είναι επίσης απόλυτα σαφές ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές, κυρίως όσον αφορά τα αιτήματα. Τα αιτήματα τα οποία αποσκοπούν ε, όχι μόνο τόσο στο να βελτιώσουμε την οδηγία, όσο περισσότερο τα αιτήματά μας είναι να ε, εναρμονίσουμε τα διάφορα εργαλεία που υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι ένας στόχος της οδηγίας θα πρέπει να είναι ένα είδος ε, κινήτρων ε, να υπάρξει κάποια βελτίωση της ε, συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και να προσπαθήσουμε και να γεφυρώσουμε το χάσμα καταπολεμώντας τη φτώχεια, κυρίως όσον αφορά τις μονογονικές οικογένειες που πολλές φορές τις περισσότερες ζουν σε απόλυτη ένδυα. Εμείς καταθέσαμε σχετική τροπολογία, ακριβώς έχοντας ως στόχο να συμπεριληφθούν οι ε, επιτιδευματίες, οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες και επιχειρηματίες, ε, οι οποίοι πολύ συχνά δεν έχουν την απαραίτητη προστασία. Μιλώ για τους επιχειρηματίες. Άρα δηλαδή είναι απολύτως απαραίτητο και από αυτού συμφωνώ με τον συνάδελφο κύριο Κάζα, είναι απολύτως απαραίτητο οι επιχειρηματίες να μπορούν να εξασφαλίσουν αυτό το δικαίωμα και να μπορούν και να κάνουν χρήση αυτού. Πρέπει λοιπόν να προβλέπονται τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα επιτρέπουν στους εργοδότες να προσφέρουν σε όλους τους εργαζόμενους αυτό το δικαίωμα. Υπάρχει το θέμα των άτυπων συμβάσεων. Είναι λοιπόν δύσκολο ε, αυτές τις εξαιρέσεις ε, εργαζομένων ε, να τις ορίσουμε. Ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε λιγάκι μεταξύ μας για να δούμε λιγάκι αυτή την κατηγορία των συμβάσεων. Εγώ είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι εκτός από την εξαίρεση των μονογονεϊκών οικογενειών θα πρέπει το δικαίωμα αυτό να το χορηγούμε και σε γονείς, ανάδοχους γονείς οι οποίοι θα πρέπει γονείς αυτοί να καταβάλουν πάρα πολλές ε, προσπάθειες, ε, ε, κυρίως όταν υιοθετούν παιδιά. Άρα σε ανάδοχους γονείς και σε γονείς που έχουν υιοθετήσει παιδιά. Πρέπει να υπάρχει τροπολογία και να στηριχθεί η τροπολογία αυτή. Όσον αφορά τώρα τα ωφέλη που πρέπει να απολάβουν οι γονείς κυρίως σε περίπτωση υιοθεσίας, αυτά τα ωφελήματα θα πρέπει να προστατευτούν. Ένα άλλο επιχείρημα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει απαραίτητα να υπάρχει κάποια πλούστευση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πλουστεύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο στη χρήση του εργαλείου. Ε, θα πρέπει όσοι παρέχουν φροντίδα να μπορούν να κάνουν χρήση μιας διαδικασίας η οποία θα είναι στάνταρτη διαδικασία και απλουστευμένη. Κατά τα άλλα, ένα άλλο σημαντικό επιχείρημα είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για την ε, έμεση ε, παροχή βοήθειας ε, μέσα στην ίδια την οικογένεια. Γιατί αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη να μπορούν να επιλέξουν κατά πόσον θα απευθυνθούν σε επαγγελματίες παρέχοντες φροντίδα ή θα μπορούσαν να απευθυνθούν στην ίδια τους την οικογένεια, η οποία η οικογένεια θα μπορούσε να συνδυάσει την παροχή φροντίδα σε συγγενείς, ηλικιωμένους ή άλλους που έχουν, εν πάση περιπτώσει, ανάγκη υποστήριξης. Εγώ πιστεύω σε μια κοινωνία που αλλάζει, στο χώρο εργασίας που αλλάζει και αυτός, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί και η έννοια της εργασίας εξ αποστάσεως, ε, της εφίους εργασίας, το smart working. Πρέπει να τα διευκολύνουμε Όπου λοιπόν ε, υπάρχουν αυτές οι μορφές εργασίας ε, και εφόσον αυτές οι μορφές εργασίας ε, προστατεύονται από κατάχρηση, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και διευκολύνει την εφαρμογή τέτοιων δυνατοτήτων. Εγώ θα συνεχίσω να μιλάω για κατάλληλες ενδεδειγμένες υπηρεσίες και για την φροντίδα των μωρών. να υπάρχουν ποιοτικέ υπηρεσίες ε, τις οποίες όμως θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα εισοδηματικά στρώματα. Ως εκ τούτου οφείλουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να προσφέρουμε κίνητρα έτσι ώστε να είναι δυνατόν να διασφαλίζει το δικαίωμα αυτό. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ε, σκέψεις που έχουμε κάνει. Όπως σας είπα, να συμπεριληφθούν οι επιτιδευματίες. Είναι προφανές ότι το κύριο επιχείρημα είναι να υπάρχει υψηλό επίπεδο ποιότητας και θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από τον συνάδελφο κύριο Κάζα να μην κατεβάζει τις προδιαγραφές, να μην υποβαθμίζει το επίπεδο, να υπάρχει ένα επίπεδο ποιότητας και να έχουμε κατά νου το βέλτιστο, γιατί είμαστε σίγουροι ότι στο Συμβούλιο θα κληθεί σε να δώσει μια πολύ περίπλοκη μάχη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, λέει ναι, κυρία Μελά. Ε, δεν σας προκαλεί εντύπωση ότι εμείς ε, μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό μήκο σχήματο σχέση με τι για πολύ απλού λόγου. Η οδηγία αυτή προβλέπει ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου για του γονεί ε, και του ε, υπεύθυνου παροχή φροντίδα, ε, είτε στα παιδιά, είτε στα παιδιά με αναπηρίε ή με δυσκολίε τροποποιώντας ε, την ε, οδηγία για την μητρική ε, άδεια, έχουμε επί της ουσίας διαφωνίας, γι' αυτό και δεν έχουμε υποβάλει τροπολογίες και θέλουμε να κάνουμε μία γνωμοδότηση μειοψηφίας. Όχι επειδή η έκθεση Καζά και οι πολλές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί δεν μας αρέσουν. Υπάρχουν πάρα πολλές σωστές ε, και ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις και προτάσεις, όμως δυστυχώς δεν εντάσσονται και δεν πρέπει να εντάσσονται σε μια νομοθετική πρόταση που υποβάλλεται προς τα κράτη-μέλη. Το ίδιο έχουμε κάνει και με όλους τους τελευταίους νομοθετικούς φακέλους που έχουν υποβληθεί και εντάσσονται στον υποτιθέμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα Δικαιωμάτων. Ε, δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά την ε, κυριαρχία των κρατών μελών, γιατί μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να καθορίσουν ε, και τον ρόλο του κράτους ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και από την άλλη τον ρόλο προσδιορίζει και τον ρόλο που πρέπει να ε, και τα δικαιώματα πρέπει να παρέχονται στους άντρες, στις γυναίκες και στους εργαζόμενους για να μπορούν να ωφελούνται διαφορών διατάξεων. Βλέπω ότι σιγά σιγά έχουμε διασχίσει μια κόκκινη γραμμή, ενώ μας μιλάτε για ισορροπία μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού βίου, βλέπουμε ότι δημιουργείται μια ανισορροπία όπου η προσωπική ζωή παίρνει το πάνω χέρι σχέση με την επαγγελματική. Καταλαώ ότι η φτωχοποίηση, τα, οι χαμηλοί μισθοί που κοντεύουν να φτάσουν στο ρόλο της φτώχειας, ε, δημιουργούν αρνητικά φαινόμενα και ότι αυτό ε, δημιουργεί δυσκολίες και στην οικογενειακό βίο και αυτό φαίνεται και από την αύξηση της παραβατικότητας και εγκληματικότητα στου νέους. Από την άλλη θέτει σε κίνδυνο και ε, όλα τα προβλήματα και όλη την δραστηριότητα των ε, επαγγελματιών, γιατί βεβαίω και ο εργοδότη δεν μπορεί να πάρει, να λάβει υπόψη όλε τι δυσκολίε που έχει ο εργαζόμενο στην προσωπική του ζωή. Και από την άλλη έχουμε και τα της ψηφιοποίησης, αυτοματοποίησης ε, και μεταστροφής της κοινωνίας και αυτό θα οδηγήσει σε τροποποίηση των ε, θέσεων απασχόλησης και θα οδηγηθούμε προς την επισφαλή εργασία. Πώς θα καταφέρουμε λοιπόν να προσαρμόσουμε τα ασφαλιστικά μας ε, συστήματα και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει ε, βιώσιμο τέτοιο σύστημα στο μέλλον εφόσον υπάρχει και ε, πτώση της κατανάλωσης ε, λόγω της πιθανής φτωχοποίησης του πληθυσμού και από την άλλη έχουμε και, τους, ε, και περιορισμό των φόρων καθώς δεν θα έχει χρήματα ο κόσμος να πληρώσει ούτε την κατανάλωση ούτε την φορολογία του για να καλυφθεί το ασφαλιστικό σύστημα και το σύστημα γενικής προστασίας ακούσουμε λοιπόν ενδιαφέρουσε σκέψεις από τις πολιτικές ομάδες, αλλά πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να θέσουν το πλαίσιο. Να αφήσουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν αυτή την άγουσα. Εμείς βεβαίω συμμετέχουμε ως κοιόδης, αλλά νομίζω ότι έχουμε περάσει αυτή την κόκκινη γραμμή και έχουμε επέμβει ε, στα χωράφια των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Κύριε Λόπες Φωτανιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν αρχίσω να ευχαριστήσω τον Ντέιβιτ για τη δουλειά του. Είναι μια πολύ καλή αφετηρία τόσο ώστε να φτάσουμε ε, σε κάποιο είδους ε, άδειε που να βοηθούν την ε, οικογενική ζωή και πιστεύω ότι όλα αυτά θα τα εγκρίνουμε πριν το τέλος της θητείας μας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για όλους τους Ευρωπαίους και αυτό θα ωφελήσει όλο τον κόσμο. Για να σταθώ τώρα σε κάποια σημεία που μου φαίνονται σημαντικά. Εάν θέλουμε περισσότερη ισορροπία μεταξύ ε, των ε, συγγενών μεταξύ των γονέων θα πρέπει πρώτα πρώτα να καλύψουμε τους ε, άντρες να είμαστε ρεαλιστές και οι οικονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να καλυφθούν από τα κράτη-μέλη, θα πρέπει επίσης μακροπρόθεσμα όλα αυτά να είναι οικονομικά βιώσιμα, γιατί δεν ωφελεί να είμαστε φιλόδοξοι αν ε, θεσπίζουμε πράγματα ανεφάρμοστα. Ε, ε, αυτό είναι ένας ρίσκος ρεαλιστικός. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει έγκριση της πρότασης και θα πρέπει όμως να πιάσει τόπο η πρόταση, δηλαδή να την εκμεταλλεύονται οι ε, άντρες. Επομένως να ρυθμιστεί και το θέμα του επιδόματος ε, και επίσης το θέμα της ε, διάρκειας. Να έχουμε επομένως μια κάλυψη 80% σε σχέση με την άδεια ασθενείας και να έχουμε με βαθμία ρύθμιση το, τη διάρκεια των 8 εβδομάδων. Οπότε να είναι ελκυστικό ο θεσμό αυτό από του άντρε και επίση να μπορεί να καλυφθεί το οικονομικό βάρο που συνεπάγεται αυτή η πρόταση. Όπω έλεγα στην αρχή, ελπίζω ότι μέχρι το τέλο τη θητεία θα μπορέσουμε να έχουμε εγκρίνει αυτή την πρόταση και έτσι θα έχουμε στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμεί εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλε τι οικογένειε. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μαγασάχτιε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αρχικά να ευχαριστήσω τον David Κάσα για ε, όλα όσα έχει κάνει και για τον τρόπο με τον οποίο εμβαθύνει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγματι θεωρώ ότι είναι ευρωπαϊκή ευθύνη και αρμοδιότητα να δείξει το σωστό δρόμο στο σύνολο των κρατών μελών. Δεν είναι θέμα επικουρικότητας, ε, είναι πραγματικά δικός μας ρόλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να εξισορροπήσουμε ε, τον επαγγελματικό και τον προσωπικό βίο και να δείξουμε στα κρατη ότι θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Το πρώτο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε και να λάβουμε δράση και αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, είναι να δοθεί τέλος ε, στην φορητότητα του, της γονικής άδειας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 2% των ανδρών μόνο παίρνουν ε, γονική άδεια. Βλέπετε λοιπόν ότι όλο το βάρος της ε, γονικής άδειας, ε, το πλεονέκτημα αυτό δηλαδή, γίνεται μειονέκτημα για τις γυναίκες, γιατί η γονική άδεια απομακρύνει τις γυναίκες από την εργασία τους, επιβραδύνει τη σταδιοδρομία τους και από τις καλές προθέσεις περνάμε τελικά στην κακή υλοποίηση. Για μένα λοιπόν το ζήτημα της μη φορητότητας του δικαιώματος είναι κέρια σημασίας γιατί αυτό είναι που θα αυξήσει ή θα γεφυρώσει το χάσμα. Δεύτερον, η χρηματοδότηση. Ακούω και σε ένα κράτος μέλος που γνωρίζω καλά φωνές που ακούγονται και θα ακουστούν και στο Συμβούλιο για το κόστος ε, του μέτρου αυτού. Όμως, εάν εξετάσουμε το ζήτημα σε, όλο, όλη του την έκταση σήμερα ε, το 60% των πτυχιούχων είναι γυναίκες. Στη σύνταξη, στην ηλικία, στην ηλικία της σύνταξης, οι γυναίκες ε, έχουν απολαβές κατά 31% χαμηλότερες. Αυτό σημαίνει ότι και τα κράτη-μέλη και οι οικογένειες επενδύουν χρήματα, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, στην μόρφωση των γυναικών, εφόσον είναι η πλειοψηφία των πτυχιούχων, αλλά στο τέλος δεν έχουμε λάβει αντίστοιχα, δεν έχει γίνει απόσβεση, αν θέλετε, αυτής της ε, ε, επένδυσης που έχει γίνει στην εκπαίδευσή τους. Ακριβώς γιατί οι εγκυμοσύνες και οι γένες αποτελούν πολύ σημαντικό πρόσκομα στη σταδιοδρομία των γυναικών. Αυτό οδηγεί στη φτωχοποίηση των γυναικών που ε, γίνεται πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα και αν ε, προσθέσετε και την δημόσια και ιδιωτική επένδυση που έγινε στην αρχή αλλά και την στήριξη που πρέπει να δώσουμε σε αυτές τις φτωχές γυναίκες κατανοείτε ότι το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο ε, την, ε, το κόστος της γονικής άδεια, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη και το κόστος που υπάρχει στην αντίθετη περίπτωση της φτωχοποίηση των γυναικών και τη εκπαίδευση που γίνεται. Και εκεί λοιπόν ε, καταλήγουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα. Ευχαριστούμε. Κυρία Ιονγκέριος έχει το λόγο. Δεν ξέρω τι να πω μετά από αυτή την ε, καταπληκτική παρέμβαση της προλαλήσας σας. Δεν θέλω να μπω στην ουσία του φακέλου, γιατί νομίζω ότι και η Μαρία Ρένα και η Ελίζαβεθ ε, τα είπαν πολύ καλά. Ήθελα μόνο εδώ να εκφράσω τη στήριξή μου ε, προς τον εισηγητή και όπως έχουν ήδη πει πολλοί συνάδελφοι προηγουμένως, είναι σημαντικό να κλείσει ο φάκελος κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θετίας. Ε, δεν θα είναι απλώς ε, αυτός ο τριμερής διάλογος, γιατί ακούμε διάφορα από το Συμβούλιο. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτή τη στιγμή να υπάρξει σαφής κοινοβουλευτική θέση και είμαι σίγουρη ότι οι εισηγητής και οι θα καταλήξουν σε ένα ε, ισορροπημένο και δίκαιο κείμενο σε μια σωστή θέση του Κοινοβουλίου. Κάτι που θα χρειαστούμε, γιατί δεν είναι απλές οι διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Να γνωρίζετε όμως ότι έχετε την αμέριστη στήριξή μας. Προχωρήστε λοιπόν και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κλείσουν αυτές τις πραγματεύσεις σε αυτή τη θητεία. Ο κύριος Γκέρνικε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Ντέιβιτ Κάζα, γιατί πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι απολύτως απαραίτητο. Ε, δείχνει ότι το όλο θέμα βράζει και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε βρει κάποια λύση. Βεβαίω ε, και πρόκειται εδώ και για την κυριαρχία των κρατών μελών. Αυτό είναι διαμφισβήτητο. Ω εκ τούτου ε, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Δηλαδή να εντοπίσουμε πού ακριβώ βρίσκονται οι βέλτιστες λύσεις ε, οι οποίες συνδυάζουν και την ε, επαγγελματική ζωή και τη φροντίδα για τους ε, οικείους. Εγώ θεωρώ ότι εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα ποσό το οποίο κατ' ουσίαν δεν μπορεί να καλυφθεί. Δεν είναι θέμα ποσού. Ό,τι ποσό και αν είναι, ε, πραγματικά πρέπει να διατίθεται. Κανένα ποσό δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτούς που προσφέρουν τη φροντίδα. Αν μιλάμε για χαρτζηλίκη τόσο μικρό δηλαδή ποσό, δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουμε. Οι γονείς και οι υπόλοιποι εκεί εξακολουθούν να είναι εξαρτημένοι και να παραμένουν οικέτες. Ναι, μεν έχουν προσφέρει πολλά στην κοινωνία, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται στο ρόλο του οικέτη. Και αυτό δεν βοηθάει στο να υπάρχει κάποια αυτοπεποίθηση στο χώρο εργασίας. Ε, εγώ ομιλώ για κάποιο ειδικό μισθό που θα ξεκινάει από μικρή ηλικία, από την ηλικία που τα παιδιά πάνε στο βερφανιπιακό σταθμό και φτάνει και μέχρι το δημοτικό. Τώρα το ότι υπάρχουν διαφορετικά ποσά, ανάλογα με το αν είμαι στη Ρουμανία, τη Σουηδία, την Αυστρία ή την Ισπανία, αυτό είναι απόλυτα σαφέ. Ω εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένας ενιαίο, ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ποσό, ε, αλλά και στην περίπτωση παροχή ε, φροντίδα ε, στου οικείου. Να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την έξω νοσοκομιακή περίθαλψη. Αυτό να είναι ο οδηγό, το οδηγό νήμα, που και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσει ακριβώ και στη φροντίδα των ε, μικρών παιδιών. Ε, τι κάνουμε. Πολύ συχνά καταδικάζουμε τις ε, γυναίκες να παρμένουν στο σπίτι, στην κουζίνα Τη στιγμή όμως που θα έχουμε ένα μισθό και θα είναι αυτός ο μισθός για την ανατροφή των παιδιών, αυτό δεν θα εξαρτάται από τους εργοδότες, θα είναι επίδομα ε, το οποίο θα καταβάλλεται από τους φόρους των φορολογουμένων με αυτό το μισθό ανατροφής τότε οι γονείς θα μπορούν να διαλέξουν αν θα παραμείνουν σπίτι να φροντίζουν τα παιδιά, να φροντίζουν τα παιδιά τους ή αν θα συνεχίσουν να εργάζονται εκτός σπιτιού. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα επιλογής και πολύ συχνά οι γυναίκες όπως ε, σας είπα συνεχίζουν να δουλεύουν για να μπορούν να καλύψουν τα προστοζήν. Υπάρχει και κάτι άλλο. Διαπιστώσαμε ότι οι γονείς καταβάλουν για τα παιδιά τους φόρους με τη μορφή του ΦΠΑ, όχι φόρο εισοδήματος, αλλά ας πούμε φόρο επί του ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, αν τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όσον αφορά τη φορολόγηση όσων έχουν παιδιά με εκείνους που δεν έχουν. Αυτό στη Γερμανία, ξέρετε, το συζητάνε ευρέως ότι είμαστε σε μια κοινωνία που όλο και περισσότερο γυράσκει ε, και να υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει κανείς αν θα κάνει οικογένεια ή όχι. Οι γονείς, όσοι δηλαδή έχουν παιδιά πολλές φορές ε, συνυπολογίζονται σε μια ειδική κατηγορία ψηφοφόρων και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αν λοιπόν αποφασίσουμε να καταβάλουμε αυτό το μισθό ανατροφής, όπως τον αποκαλούμε, θα υπάρχει μια μορφή δικαιοσύνης. Θα μπορεί κανείς να συγκρίνει ε, αυτούς που έχουν παιδιά με τους άτεκνους και Μόνο σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι θα μπορούμε να καταλήξουμε και σε μια πιο δίκαιη σύνταξη. Γιατί όσον αφορά τον υπολογισμό των συντάξιμων ετών ε, θα πρέπει να συνυπολογίζονται τα χρόνια ανατροφής. Όχι με τη μορφή χαρτζηλικιού αλλά με τη μορφή μισθού. Και εγώ εδώ ε, θεωρώ ότι έτσι θα υπάρχει ε, δικαιοσύνη πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη σύμβαση ανάμεσα σε δύο γενιές, να πάμε σε μια άλλη μορφή, σε σύμβαση, σύμβαση τριών γενεών. Γιατί όπως και οι συνταξιούχοι και τα παιδιά δεν κερδίζουν χρήματα και πρέπει να χρηματοδοτούνται. Ως εκ τούτου, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει, εφόσον θέλουμε δικαιοσύνη στο θέμα των συντάξεων, νομίζω ότι πρέπει να δείτε λιγάκι το θέμα των γυναικών και θα διαπιστώσουμε ότι κυρίως οι γυναίκες πλήττονται από την ε, φτώχεια στην τρίτη ηλικία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες, να διεκδικήσουμε μια Ευρώπη η οποία μακροπρόθεσμα δεν θα είναι μια γυρασμένη κοινωνία. <coughs> Γιατί διατρέχουμε αυτή τη στιγμή αυτόν τον κίνδυνο να αδειάσουν τα κοινωνικά μας ταμεία. Κύριε Κάζα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνδυάζετε για τους γονείς, η οικογένεια με την εργασία. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Ε, δεν ξέρω αν ο εισηγητή θέλει να ολοκληρώσει αυτό το θέμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα με γρηγορήσω γιατί ξέρω ότι πιεζόμαστε χρονικά. Ε, πάντως ε, νομίζω ότι όλος ο συνάδελφοι σε αυτή την με στη συζήτηση ήταν πολύ σημαντικά και θα πρέπει να σας πω και πάλι αυτό που σας είπα στην αρχή νομίζω πως είναι σημαντικό το εξής να καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό αλλά να μην υπερβάλλουμε προς ε, το ένα ή το άλλο άκρο να προσπαθήσουμε να βρούμε τη μέση οδό να καταλήξουμε σε κάτι ισορροπημένο, σε κάτι εφαρμόσιμο και πρακτικό. Να μην πάμε στο Συμβούλιο με θέσεις που δεν επιδέχονται συμβασμούς μαζί τους. Άρα ως Κοινοβούλιο να καταλήξουμε σε ε, μια τελική θέση και να πάμε έτσι στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Σας είπα, δεν θεωρώ πρόβλημα το να συνοηθούμε μεταξύ μας. Πάντως να ευχαριστήσω και πάλι τους και ιδέες. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες, θα βρούμε ε, κάποιες συμβαστικές διατάξεις και θα μπορέσουμε έτσι να βρούμε μια λύση ή ισορροπημένη πρόεδρος. Ευχαριστώ και τον κύριο Κάσα και όλους τους αδελφούς οι οποίοι συμμετέσχουν στην συζήτηση. Ε, νομίζω τα πράγματα ξεκαθαρίστηκαν, το τι, τι πρεσβεύει ο καθένα. 11 Ιουλίου θα εγκρίνουμε το κείμενο, δηλαδή την τελευταία μα συνεδρίαση πριν τις θερινές διακοπές. Τουλάχιστον για μας από την Βόρεια Ευρώπη. Άρα επανερχόμαστε στο θέμα. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης. Πρόκειται για την αύξηση του κονδυλίου για το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Προσαρμογή του γενικού στόχου. Δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσάμπα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως τα γνωρίζετε, αυτό το πρόγραμμα καθορίστηκε πέρσι για την περίοδο 17 με 20 για 142,8 εκατομμύρια, ούτως ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τις μεταρρυθμίσεις και να έχουν την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν ζητήσει οι κυβερνήσεις. Οπότε είπαμε ότι έχουμε κάποιους τομείς ε, σημαντικούς όπως κατάρτιση, εκπαίδευση, ε, αγορά απασχόλησης, ε, θέσεις απασχόλησης, καταπολέμηση της ε, φτώχειας, κοινωνική ένταξη, κοινωνική πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση, δημόσια υγεία και επίσης και για άλλους τομείς που έχουν σημασία για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Πρώτα-πρώτα για αυτό το πρόγραμμα το 17 και το 18 ήταν πολύ θετικά τα κράτη-μέλη και φτάσαμε σε 152 εκατομμύρια ευρώ ε, ως αίτημα, πέντε φορές δηλαδή παραπάνω από το αρχικό κονδύλι και ε, πάμε ότι αυτό είναι λογικό και έχουμε επίσης κάποιες άλλες δεσμεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρητά προβλέπει ότι θα πρέπει Εξαστεί ποια κράτη-μέλη θέλουν να μπουν στην Ευρωζώνη. Τώρα, προσπάθησα να καλύψω τον στόχο του να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη για τις προσπάθειές τους να μπουν στην Ευρωζώνη. Είναι στόχος του προγράμματος. Και επίσης το πρόγραμμα αυτό, SRSP, να είναι δυνατότητα για όλα τα κράτη-μέλη και για τα μέλη της Ευρωζώνης και για τους άλλους. Επίσης θέλω να τονιστεί το ότι χρειάζονται διορθικές μεταρρυθμίσεις για τις κοινωνικές πολιτικές και να καλυφθεί η ανάγκη για παραγωγικότητα, για επαγγελματική κατάρτιση και ενεργή πολιτική επασχόληση. Πολύ σημαντικό αυτό να ε, λάβουμε υπόψη ότι σήμερα Έχουμε τους στόχους για την απασχόληση το 2020 για την γενική ένταξη, στόχοι που ε, ακόμη δεν έχουν επιτευχθεί. Είναι κατακλείδη πολλά κράτη-μέλη δυσκολεύονται για το πώς θα εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Και η Ουγγαρία πρόσφατα έκανε κάποιες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων αλλά πάρα πολύ δεν καλύπτουν αυτέ τι μεταρρυθμίσει, ιδίω στον τομέα τη υγεία και είναι τώρα σε χειρότερη θέση. Οπότε μπορεί αυτό το πρόγραμμα να βοηθήσει. Πρόκειται μια προσπάθεια από την βάση να βελτιωθούν οι διοικητικέ δυνατότητε και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη απορρόφηση των κοινωνικών κονδυλίων. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι πρόσφατα το Συμβούλιο συμφώνησε να αυξήσει την προεκοδότηση. Και επίσης Έχουμε τα αρχικά αποτελέσματα που οδήγησαν στην Επιτροπή να δώσει 25 ε, δις για την επόμενη δημοσιονομική χρήση. Πώς βλέπω στην συνεργασία με τους σκιώδεις συζητητές και παρακαλώ οι συνάδελφοι να υποβάλουν τις τροπολογίες στα αγγλικά για να μπορέσουμε εγκαίρως να ολοκληρώσουμε τη γνωμοδότησή μας και να τις υποβάλουμε στην κυρίως αρμοδία επιτροπή. Ευχαριστούμε που αναφέρατε και την προθεσμία κατάθεση τροπολογίων 22 Μαΐου. Και επειδή είναι τόσο λίγος ο χρόνος, καλέσατε κατά τη μελη να υποβάλουν τις τροπολογίες τους στα αγγλικά για να μπορέσουν να περιληφθούν στις συμβαστικές. Δεν είναι υποχρέωση αυτό, απλώς ε, θα απλοποιούσε τα πράγματα. Ο κύριος Περίνσκι τώρα, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Σόγκορ, για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, που μας παρουσίασε. Νομίζω ότι καλύπτει ε, τα βασικά στοιχεία της θέσης που πρέπει να έχει η Επιτροπή μας σε αυτό το ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα συμμερίζουμε την άποψή του ότι η χρήση στρατηγικών προτεραιοτήτων ε, στην ετήσια έκθεση προόδου είναι σημαντική σε τομείς όπως η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η παραγωγικότητα ε, της αγοράς, στην αγορά εργασία και η κοινωνική συμπερίληψη. Θα πρέπει να υπογραμμιστούν περαιτέρω όλα αυτά στο πλαίσιο ε, της υλοποίηση του προγράμματος στήριξης διαθετικών μεταρρυθμίσεων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την υλοποίηση νέας γενιάς διαθετικών μεταρρυθμίσεων που πλέον από τη λιτότητα θα περνάει σε μία εξισορροπημένο συνδυασμό ε, διαφόρων ε, μέσων για να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη για όλα τα κρατημέλη. Έχουμε και τα αποτελέσματα του του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για όλα τα κρατη και βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι βίωνα. Σε πολλές χώρες τα πράγματα είναι κρίσιμα. Για τουλάχιστον έναν από τους 12 ε, δείκτες, δύο χώρες είναι σε κρίσιμη κατάσταση για έξι δείκτες, η Βουλγαρία είναι για πέντε. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ανισότητα εισοδημάτων, ε, τον κοινωνικό αποκλεισμό και ούτε καθεξής. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι διορθωτικέ μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα δεν έχουν φέρει αυτή τη ε, μεταμόρφωση που ε, να διασφαλίσει ε, μια αξιοπρεπή διαβίωση για τους Ευρωπαίους πολίτες. Επομένω, οι μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στους οικονομικούς δείκτες αλλά και στη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και το καθεξής. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος που προανέφερα, όμως τα συνοπτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή ΡΕΤΖΙ το Φεβρουάριο, τα παρουσίασε ο Επίτροπος Δομπρόφσκης, δείχνουν ότι το 27% το, η μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης για το 2017 κατανεμήθηκε στον τομέα πολιτικής της αγοράς εργασίας, τη υγεία και των κοινωνικών υπηρεσιών. Για το 2018 το μερίδιο για αυτό τον τομέα πολιτικής είναι 21%. Υπήρξε πολύ σημαντικό αριθμό αιτήσεων για το 2017 και το 2018. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον από τα κράτη-μέλη και το σημαντικό μερίδιο τη χρηματοδότηση που δίνεται για τον τομέα της κοινωνική αγοράς ε, και της πρόνοιας δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη θέλουν βοήθεια. Η αύξηση λοιπόν μπορεί να στηριχθεί, όμως ε, υπογραμμίζοντας ότι οι πόροι θα πρέπει να προκύψουν από τον, ε, το μηχανισμό ευελιξίας υπό τον επόμενο ΠΔΠ και όχι σε βάρος άλλων πολιτικών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει η τροπολογία στον υφιστάμενο κανονισμό που να επισημαίνει ακριβώς αυτό. Άλλη πρόταση για να αναφέρουμε ρητό στη συμβολή του προγράμματος για τη στήριξη προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων για, την ένταξη των κρατών μελών στην Ευρωζώνη υπενθυμίζουμε ότι και στα υφιστάμενα προγράμματα υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Η Επιτροπή προτείνει νέο μηχανισμό υπό το επόμενο πιδελταπή, συμπερίληψη ξεχωριστού στόχου για την στήριξη στην προετοιμασία της ένταξης στην Ευρωζώνη φαίνεται σε μια δοκιμαστική φάση αυτής της πρότασης και γύρει νέα αιτήματα για την πρακτική χρησιμότητα του μέσου αυτού. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα νέο μέσο, το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά το 2020, καθώς σε υλοποίηση του προγράμματος βρίσκεται στην αρχική φάση, δεν υπάρχουν στοιχεία για το πραγματικό αντίκτυπο και προσθεμένη αξία που θα έχει. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή να μας δίνει τακτικά πληροφορίες για την εφαρμογή. Ο κανονισμός 2017 κάθετος 825 αναφέρει στο άρθρο 16 ότι η Επιτροπή ετησίως θα υποβάλει έκθεση παρακολούθησης για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά δεν προσδιορίζει το έτος έναρξης και λήξης για την υποβολή των εκθέσεων. Αυτό μπορεί να διορθωθεί με σχετική τροπολογία στο άρθρο 16. Και εγώ, κυρία Πρόεδρε, προσβλέπω σε συνέχιση συνεργασίες με τον εισηγήτη και τους κοιότητες και αυτό θα ευχαριστώ. you, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Πυρίνσκι. Από το ECR δεν βλέπω κάποιον. Ούτε από την Άλντε. Επομένως... Έχετε το λόγο κύριε Σιλικιώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που επετέλεσε. Σε κάθε περίπτωση όμως η GUEGL ε, ως QRGL πρέπει να επαλάβουν τη θέση μας ε, όταν την διατυπώσαμε και πριν 1,5 χρόνο γιατί ξανασυζητήσαμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Για μας οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επιβάλλονται στα κράτη-μέλη αλλά και η διασύνδεση των πολιτικών της ΟΝΕ με αυτές του Ευρωπαϊκού Εξαμένου δεν κινούνται στη λογική τη πρόσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων πόσο μάλλον τη πρόθεση της κοινωνική συνοχή. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε να γίνεται είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ πλουσιών και φτωχών, η διάλυση του κοινωνικού κράτους, η παγωποίηση των ψηλών ποσοστών υγεία και φτώχεια στην εργασία. Αυτές ε, για μας είναι οι καταστροφικές επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται μέσα από την ΕΕ και των Ευρωπαϊκών και πρέπει να σα πω ότι ε, σε αρκετές χώρες οι εργαζόμενοι κυρίως στην περιφέρεια, ε, ε, βίωσαν με βίαιον τρόπο, μέσω των μνημονίων, αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις βιώνουν ακόμα ε, και οι εργαζόμενοι στο σκληρό πυρήνα του ευρώ. Δεν αρκούν οι θυσίε των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια ως δίθεν λύση για την οικονομική κρίση. Η, η Κομισιόν, το Συμβούλιο και οι, οι Τρόικες που εγκαθίδρανται σε διάφορες χώρες προωθούν ακριβώ τέτοιου μηχανισμού που κατά την άποψή μα και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα διευρύνουν τι ανισότητε. Ε, σε αυτό το πλαίσιο θα καταθέσουμε και φέτο όπω και την προηγούμενη φορά τροπολογίε στο πνεύμα που ανάφερα πιο πάνω οι οποίε πρωτα πρώτα-πρώτα να υπογραμμίζουν τι αρνητικέ συνέπειε αυτού του λεγόμενου δημοσιονομικού συντονισμού. Επίση, θα τονίσουμε την ανάγκη ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτου, τη κοινωνική συνοχή τη δημιουργία νέων αξιοπρεπών θέσεων εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώματα μέσω δημόσιων και μακροχρόνων επενδύσεων. Βεβαίω, παράλληλα, πρέπει να σημειώσω και να χαιρετήσω την τροπολογία νέα του εισηγητή για την εισαγωγή του άρθρου 9 και 11 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Οδηγία, αλλά και κάποιε αναφορέ για δυνάμωση των κοινωνικών πολιτικών, όπω αναφέρονται για παράδειγμα στι τροπολογίε 3, 4 και 8. Εν τούτης, εμείς έχουμε σοβαρούς ευθυασμούς όσον αφορά ε, την τροπολογία 6, η οποία καλεί για πόρους στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα αφορούν μόνο ε, τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, και όχι βεβαίως τις κοινωνικές πολιτικές. Παρά τις διαφορίες μας με το πνεύμα της νομοδότησης και της οδηγίας, εμείς θα συμμετέχουμε στη συναντήση των σκηνών εισηγητών με επικοδοτικό πνεύμα και θα καταθέσουμε, όπως ανάφερα, ε, τις δικές μας τροπολογίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο και πάλι στον κύριο Σόγκορ, αν ε, θέλει να δευτερολογήσει. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τις παρεμβάσεις σας. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 22 Μαΐου και καλείστε να τις υποβάλλετε στα αγγλικά για να συμπεριληφθούν ε, στις συμβαστικές τροπολογίες. Ε, στην Επιτροπή μας θα ψηφιστεί πρώτα στις 7 Ιουνίου και στη Ρέτζη ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί η ημερομηνία. Έχουμε φτάσει στο τέλος της μέσης διάταξης. Διακόπτουμε εδώ λοιπόν και επιστρέφουμε στις 2.30 για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Α, ο κύριος Πυρίνσκι πρώτα. Ε, βλέπω ότι έχετε και ένα άλλο σημείο εδώ, υπό τα διάφορα. Μπορούμε να αφιερώσουμε ένα λεπτό. Ναι, λέει η Πρόεδρος, φυσικά έπρεπε να το είχα αναφέρει και εγώ ε, υπό το 8. Παρακαλώ κύριε Πρίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με τον έλεγχο ε, των οδηγών στα οδικά δίκτυα, ιδίως στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Γιατί υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες ε, προκύπτουν από τους ελέγχους των οδηγών. Και ένας Ρουμάνος οδηγός θέτει αυτό το ζήτημα ε, σε πολλούς ευρωβουλευτές, γιατί αυτή τη στιγμή οι ελεγκτικές αρχές ζητούν αποδεικτικά στοιχεία για την προϋπόθεση, για τον κανόνα που υπάρχει, που ακόμα δεν έχει νομοθετηθεί, η τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα, ανάλογα πώς μετράει κανένας, να την περνάει σπίτι του. Να είναι αυτή η ανάπαυση. Παρότι οι οδηγοί έχουν αποδείξει ότι πέρασαν αυτή την εβδομάδα ανάπαυσης εκτός του οχήματος έχουν ε, ε, λάβει τεράστια πρόστιμα, χιλίων και δύο χιλιάδων ευρώ, που πραγματικά είναι κάτι απαράδεκτο και υπάρχουν σημαντικές συνστάσεις, εφόσον ακόμα δεν έχει καν περάσει αυτή η νομοθεσία. Βρίσκεται σε μορφή προσχεδίου. Εγώ λοιπόν θα μεταφέρω αυτό το, το μήνυμα ε, του Ρουμάνου οδηγού το θέτω υπόψη σας και των συναδέλφων στην Επιτροπή Απασχόλησης και ελπίζω να λάβουμε ξεκάθαρη θέση κατά τέτοιων αυθαίρετων ελέγχων χωρίς νομική βάση οι οποίοι εφαρμόζονται πολύ επιλεκτικά κατά ε, των οδηγών από ορισμένε ε, ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Ήθελα απλώς να τα επισημάνω. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση. Θα το διερευνήσουμε. Ίσως και η Επιτροπή Μεταφορών ε, να μπορεί να επιληφθεί ή ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερωθούν τουλάχιστον για την υπόθεση. Οπότε πρέπει να βρούμε περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες και θα επανέλθουμε. Ιδάλλως θα μας το επενθυμίσετε. Σας ευχαριστώ τα ξαναλέμε στις 2.30 και μισή στις ψηφοφορίες. Thank you for this, uh, morning